Buongiorno a tutti, vi prego. Καλημέρα σα, σα παρακαλώ καθίστε. Buongiorno, cominciamo la... Να ξεκινήσουμε με τη συνεδρίασή μας. ήθελα να προσέξετε τώρα για ορισμένε ανακοινώσει. Από τη στιγμή που ορισμένε πολιτικέ ομάδε ε, δεν κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν τι διαβουλεύσει του, το σημείο 4 που αφορά την εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου. Το σημείο αυτό θα το δούμε λοιπόν στην επόμενη συνεδρία, στο να βάλουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τη σημερινή ημερησία διάταξη, το σχέδιο σας προτείνω μια τροποποίηση. Είχαμε σκεφτεί πρώτα να έχουμε παρουσίαση του συγχητή κατόπιν ε, τη συζήτηση και κατόπιν παρουσίαση των εκθέσεων των άλλων δύο συναδέλφων ε, του κυρίου Μποριέτσε και του κυρίου Ταβάρες. Αυτό λέει στην δημοσία διάταξη. Εγώ όμως θα σας πρότεινα να ακούσουμε όλους τους συντάκτες των εγγράφων και κατόπιν να περάσουμε στη συζήτηση. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, προτείνω να εγκρίνουμε τη μερσία διάταξη έτσι όπως ε, τροποποιήθηκε και σας ανακοινώθηκε. Μάλιστα, περνάμε στο σημείο 2 αν δεν υπάρχουν παρατηρήσει ή αντιρρήσει, να εγκρίνουμε τα πρακτικά τη συνεδρίασης τη 23 και 24, 23, Ιανουαρίου 2013, έτσι όπω έχουν σταλεί. Να περάσουμε στι ανακοινώσει τη Προέδρου. Έχω δύο ανακοινώσει. Ο Πρέφη Λαφατόνσοφ από τη Βουλγαρία προσχώρησε στην Επιτροπή μα και αντικαθιστά την Ιλιάνα Ιβάνοβα από τη Βουλγαρία, ο κύριος Σαλβατόρε Καρόνα ε, και αυτός προσχώρησε στην ΚΡΙΜ ε, από την ομάδα των σοσιαλιστών ως τακτικό μέλος. Και ε, να σας πω ότι στη συνεδρίαση αυτή αναμεταδίδεται και μέσω του διαδικτύου και να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα αυτή θα έχουμε και τη συνεδρίαση των συντονιστών της ΚΡΙΜ στις 5.30. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην ουσία. Όπως όλοι γνωρίζετε, η εντολή της Επιτροπής μας προβλέπει την παρουσίαση μιας ενδιάμεσης και μια τελικής έκθεσης. Ο κύριος Γιακολίρο είναι ο εισηγητής και σήμερα θα μας παρουσιάσει ορισμένες πτυχές θα παρουσιάσει τρία διαφορετικά έγγραφα που έχουν να κάνουν με το οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και την νομιμίωση υπό όρων από παράνομες δραστηριότητες. Ε, ο εισηγητής σε σχέση με το τρίτο έγγραφο εργασίας ε, βάσει και των δημόσιων ακριώσεων που θα γίνουν και βάσει διάφορων θεματικών εγγράφων που έχουν, ε, που έχουν παρουσιάσει, μάλλον έχουν συγγνώμη, συντάξει κύριοι Μποργέζε και Ταβάρες θα βασιστεί στις πληροφορίες αυτές κατόπιν ε, τώρα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γιακολίνο, κατόπιν στους κύριους Μποργέζα και Ταβάρης για 10 λεπτά και θα περάσουμε στη συνέχεια στη συζήτηση. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γιακολίνο για 20 λεπτά. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μου δίνετε αρκετό χρόνο. Θα προσπαθήσω όχι μόνο να σεβαστώ το χρόνο, αλλά και να μην μακρηγορήσω, να παρουσιάσω το περιεχόμενο αυτού του τρίτου εγγράφου εργασίας ε, πιο σύντομα. Είμαστε λοιπόν στο τρίτο εγγραφό εργασίας, ε, όπως είπατε και εσείς προλίγου. Και το ένα αφορούσε το οργανωμένο το άλλο τη διαφθορά και με τη βοήθεια των συναδέλφων και την υποστήριξη των κυρίων Ταβάρες και Μποργκές με τη συνεισφορά τους και αυτοί με βοήθησαν τα μάλα και επίσης και με τη βοήθεια της γραμματείας ε, καταλήξαμε σε αυτό το τρίτο έγγραφο εργασίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, ε, είχαμε και μία συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές στο Στρασβούργο τις εβδομάδες, ε, τις προηγούμενες, κατά τη διάρκεια της τελευταίας ε, Ολομέλειας, όπου συμμετείχαμε. Σημαντικά στοιχεία πήραμε και από τη συνεισφορά των συναδέλφων Μπορκέτζο και Ταβάρες και μάλιστα ο κύριος Μπορκέτζο μας περιέγραψε με πολύ μεγάλη ακρίβεια τη σχέση μεταξύ τραπεζών και χρηματοδότησης και επίσης πολύ σημαντική ήταν και η συσφορά του κυρίου Ταβάρε σε σχέση με θέματα που έχουν να κάνουν με τη φοροδιαφυγή, την φοροπάτη και τους φορολογικού παραδείσει και το συνολικό πλαίσιο αναφοράς που πρέπει να παρέχεται ως εγγύηση για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών οι παρατηρήσεις τους, οι παραπομπές τους και οι ιδέες τους φυσικά βρίσκουν αναγνώριση στο έγγραφο εργασίας και φυσικά εκεί αναφέρουμε ως απειλή το θέμα που έχει να κάνει με το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος και αναφέρεται πόσο μπορεί να θίξει την χρηματοοικονομική σταθερότητα και τον πλούτο της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε σημαντικές ε, πηγές που αφαιρούνται, σημαντικούς πόρους που αφαιρούνται από την νόμιμη οικονομία και πλήττουν την ευημερία των πολιτών. Έτσι καταλήγουμε σε ένα πολύ σημαντικό έγγραφο που έχει να κάνει και με την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. Υπολογίζουμε ότι το περασμένο έτος ε, ένα δισεκατομμύριο 600 εκατομμύρια δολάρια είναι ο αριθμός ε, το ποσού που ξεπλήθηκε παγκοσμίως. Ε, μιλάμε στο 2,7 του παγκόσμιου ΑΕΚΠ. Είναι ένα σημαντικό ε, νούμερο αυτό και βλέπετε ότι το φαινόμενο αυτό είναι παρόν, υπάρχει παγκοσμίως αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα μεμονωμένα κράτη-μέλη μέσω ενός πανοράματος που φυσικά διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Τι προσπαθήσαμε τώρα εδώ να εντοπίσουμε, να προσδιορίσουμε σε αυτό το τρίτο έγγραφο. Προσπαθήσαμε να προσφέρουμε μία σαφή δομή, μία μεθοδολογία απλή και προσβάσιμη αφού ζητήσαμε από την Επιτροπή έναν ενιαίο ορισμό για την νομιμοποίηση παράδομων εσόδων και σκεφτήκαμε ότι πρέπει να βρούμε ποιες είναι οι πιο κατάλληλες τεχνικές καταπολέμησης. Επίσης, απεικονίζουμε το νομοθετικό πλαίσιο και αναφέρουμε τις καλύτερες εθνικές εμπειρίες. Επίσης προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις, ε, προσπαθήσαμε να δούμε ε, κατά πόσο υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών και των ενδιάμεσων και άλλων ε, επαγγελματικών κατηγοριών. Ε, στην Ιταλία μόνο έχουμε διπλασιασμό σε σχέση με το 2011. Το 2012 διπλασιάστηκε ο αριθμός των ύποπτων συναλλαγών κάποιες από τις οποίες έχουν διασυνοριακή φύση και θα μπορούσε από εκεί να προκύψει μια προσέγγιση που να βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου. Και βλέπουμε ότι το φαινόμενο της νομικής παρανοσόδων ε, είναι ε, παρόν στα κράτη-μέλη. Έχουμε προβλέψει ορισμένους τρόπους πρόληψης αλλά και καταπολέμησης, νέες μεθόδους πληρωμών, μία πιθανή μείωση ε, της... Ε, μάλλον μία ανιχνευσιμότητα, επίσης να προσφεύγουμε σε όσων διαδραματίζουν ένα ρόλο σε αυτές τις συναλλαγές. Ο κύριος Μποργκέτσιο μας ε, παρουσίασε ε, τι συμβαίνει με τα τυχερά παιχνίδια στο ίντερνετ, τα online τυχερά παιχνίδια, τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια και εκεί δεν υπάρχει αποτελεσματική καταπολέμηση. Υπάρχει θέμα αδειών αλλά και θέμα ελέγχου. Ανιχνευσιμότητα του χρήματος είναι μια συγκεκριμένη απέτηση. Πολύ συχνά αναφερόμαστε σε διασυνοριακές συναλλαγές και χρειάζεται εκεί ένας μηχανισμός συνεργασίας ε, και κατάδειξης ε, αυτών των συναλλαγών. Επίσης, ε, τονίσαμε, δώσαμε έμφαση στην ε, πρόβλεψη του αδικήματος του αυτοξεπλήματος, self-laundering, ε, υπάρχει ε, αυτό το αδίκημα σε ορισμένα κράτη-μέλη, ορίζεται ως τέτοιο. Ο κύριος ε, Ταβαρές αναφέρεται και στους φορολογικούς παραδείσους, σε αυτά τα φαινόμενα που είναι πάρα πολύ σοβαρά και πολύ συχνά σημαίνουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία να εντοπιστούν αυτές οι διασυνοριακές συναλλαγές. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, μεταφορές περιουσιακών στοιχείων σε φορολογικούς παραδείσους και επίσης ε, εκεί είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε αν υπάρχουν συναλλαγές που έχουν νομοποίηση παράνομων εσόδων. Χρειάζεται μεγαλύτερο έλεγχος και εποπτεία. Θέλουμε να έχουμε καλύτερη τραπεζική διακυβέρνηση, μεγαλύτερη τραπεζική διακυβέρνηση που να σημαίνει μεγαλύτερη συνεργασία και μεγαλύτερη ικανότητα παρέμβασης ε, των ελεκτικών μηχανισμών ε, θα πρέπει ο νέος μηχανισμός να ενισχυθεί με την ε, τραπεζική εποπτεία και την καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομων εισόδων ε, και εκεί ο κύριος Ταβάρες εστιάζει στο δική του θεματική συνεισφορά. Επίσης αναφερθήκαμε και στο διεθνές νομοθετικό πλαίσιο, στο ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της ε, Task Force, ε, της ΓΚΑΦΗ ε, και η σύμβαση του θα πρέπει να επικυρωθεί και να τεθεί σε εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, μιλήσαμε για τη σχέση της νομοποίησης παραμεσόδων με τα ε, καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ε, και αναφερόμαστε στο ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίσης, αναφερθήκαμε συγκεκριμένα στις συστάσεις της ΓΚΑΦΗ που προωθήθηκαν με αποφασιστικότητα. Εν μεταξύ, επίσης, αναφερθήκαμε στο ρόλο της Επιτροπής και του Συμβουλίου και συχνά εκφράσαμε την απέτηση να υπάρχει μία ομοιομορφία σε ε, ό,τι αφορά το ρόλο ε, των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών Σίγουρα μέσα από αυτές τις συγκεκριμένες δραστηριότητες μετρούμε το βαθμό της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Εν τω μεταξύ η Κομισιόν έκανε μία πρόταση οδηγίες για την καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομης οδών και σίγουρα θα έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις για το θέμα αυτό στην ε, Επιτροπή όπου θα λάβει χώρα η συζήτηση αυτή τις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε αναφερθεί σε ορισμένε εμπειρίε στην Ιταλία, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στι κάτω χώρε. Για το self learning, και το αυτοξέπλυμα υπάρχουν ε, διαφορετικέ καταστάσει. Προβλέπεται στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία αυτό το αδίκημα, ενώ σε άλλα κρατημέλη δεν προβλέπεται και θα επιθυμούσαμε να έχουμε μια ενιαία θέση σε όλα τα κρατημέλη και επίσης ε, και το ίδιο να ε, ισχύει και για το θέμα του προπολογισμού. Να έχουμε μία προσέγγιση αξιόπιστη. Συμπέρασμα, Πρόεδρε. Ο στόχος ε, σε συνεργασία με τους συντενιστές, με τους σκιώδες, με τους συναδέλφους και με την Κομισιόν, ο στόχος που έχω θέσει με ε, τη συνεχή στήριξη της Προεδρίας ε, και της Γραμματείας είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο. Δηλαδή θα πρέπει να κατεπολεμήσουμε αποτελεσματικά τη μαφία, το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά όπως και την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Να έχουμε ενιαία κριτήρια για τη στατιστική καταγραφή του φαινομένου του ξεπλήματος, να υπάρχει υποχρέωση ε, της καταγγελίας των ύποπτων συνολογών και όπως είπαμε ε, να έχουμε έναν ομοιόμορφο ρόλο των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών να υπενθυμίσουμε ότι η νομοποίηση παράνομων εισόδων ε, έχει συγκεκριμένες πτυχέ λειτουργίας που συνδέονται με την ικανότητα οργάνωση των ε, εγκληματικών συστημάτων που έχουν ε, παγκόσμια και διεθνή φύση και βεληνικέ και πρέπει να ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για να μπορούμε να ανοιχνεύουμε τι συναλλαγές. Επίσης, όπως πρότεινε και ο κύριος να προβλέψουμε την άρση της ανωνυμίας όσων παίζουν τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να έχουμε επαρκή εποπτή αυτής της δραστηριότητας, να αξιολογήσουμε τους κινδύνους που ενέχουν τα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα και να δώσουμε και ένα ρόλο στα εμπορικά επιμελητήρια προκειμένου να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους έντιμους εμπόρους, αλλά και να ποινικοποιήσουμε όσους δεν είναι έντιμοι. Επίσης, έχουμε προβλέψει οι επιχειρήσεις που έχουν καταδικαστεί ε, για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος να μην μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες ε, δημοσίων συμβάσεων, ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Όποιος έχει καταδικαστεί για νομιμοποίηση παράδομων εισόδων σε ένα κράτο μέλος να μην μπορεί να συμμετάσχει σε διαδικασίες ε, ε, ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ούτε και σε άλλα κράτη-μέλη για να προστατεύσουμε τους τίμιους εμπόρους. Επίσης προβλέπουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις ε, για, την, ε, ε, για μέτρα κατά της πολέμησης του, της παράνομων εσόδων για να προστατεύσουμε τι εμπορούς Επίσης, δέουσα επιμέλεια για τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ένα ρόλο εποπτείας στις τραπεζικές αρχές που έχουν αυτό το ρόλο όπως προβλέπεται από την κοινωτική νομοθεσία προοδευτική αξιολόγηση του ρόλου που η Τραπεζική Ένωση στην Ευρώπη θα μπορούσε να διαδραματίσει μεγαλύτερη διακυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα φορολογικά. Πρέπει να δούμε το θέμα της φορολογικής απάτης που σχετίζεται με τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Ε, δεν έχει να κάνει μόνο με τις περιοχές σύγκλησης αυτό. Επίσης περισσότερος έλεγχος, καλύτερη ενημέρωση ε, και καλύτερη κατάρτιση των αστυνομικών και των, και των δικαστών. Επίσης ε, πρέπει να υπάρχει και η μηβαία κατανόηση των προβλημάτων που μπορεί να εγγυηθεί στις διοκτικές αρχές τους τους δικαστές επιτυχία στις ε, δραστηριότητες τους. Και κλείνω λέγοντας ότι οι δραστηριότητες ε, που αναφέρονται καταδεικνύουν μια μεγάλη συνεργασία με τους συναδέλφους, με την Γραμματεία και με την Προεδρία. Έχουμε φτάσει σε προχωρημένο στάδιο και για την ενδιάμεση έκθεση και μέσα σε αυτή την εβδομάδα στις 22 του μήνα πιστεύουμε ότι θα ολοκληρώσουμε την ενδιάμεση έκθεση που θα κατατεθεί σε όλους εσάς και θα παρουσιαστεί στις 18 Μαρτίου. Πήρα και μια σειρά συνεισφορών από τις πολιτικές ομάδες και φυσικά θα τις χρησιμοποιήσω όταν ε, θα ολοκληρωθεί το έγγραφο που θα αποτελέσει αντικείμενο της ενδιάμεσης έκθεσης και θα παρουσιαστεί σε εσά στις 18 Μαρτίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Γιακολίνο. Από όσα ακούσαμε, κατανοούμε πώς ε, σήμερα παίρνει ζωή ο στόχος που είχαμε θέσει στην ε, έναρξη της θητείας αυτής της Επιτροπής όταν είχαμε ε, μιλήσει για τις δυσκολίες που μπορεί να ενέχει η εναρμόνιση 27 διαφορετικών συστημάτων, νομικών συστημάτων για να κατανοήσουμε το οργανωμένο έγκλημα ως απειλή, που απειλεί όχι μόνο ε, την οικονομική ζωή, αλλά απειλεί και όλο το νομικό σύστημα. Ακούσαμε λοιπόν από τον εισηγητή μας ε, κάποια πολύ ισχυρά κριτήρια. Ε, σε λίγες χώρες υπάρχει το αυτοξέπλημα ως αδίκημα, όμως θα πρέπει να ισχύει και στις 27 χώρες. η καταπολέμηση θα πρέπει να είναι χωρίς δισταγμούς, αλλά θα πρέπει να γίνει και με ίσα όπλα έναντι όλων των φορολογικών ε, παραδείσων. Φανταστείτε ότι κάποιος θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί κάποια συστήματα που δεν θα υπάρχει ο έλεγχο στον οποίο αναφερθήκατε εσεί πριν. Ε, έτσι λοιπόν ε, θα μπορούσαμε να θέσουμε το θέμα αυτό ως προτεραιότητα της δικής μας ε, θητεία μας το 2014. Γιατί η δική μας επιτροπή, το έργο μας δεν θα οδηγηθεί δεν θα οδηγήσει μόνο σε κοινούς καρπούς, αλλά εδώ έχουν παρουσιαστεί και κάποιε ιδεολογίε πολιτικών ομάδων, αλλά όλοι οι βουλευτέ και όλοι οι πολιτικέ ομάδε έχουν συμφωνήσει στο ότι είναι αναγκαίο να προσφέρουμε δημοκρατία, ελευθερία και ασφάλεια στου Ευρωπαίους πολίτε. και πρόκειται για κάποιε αρχέ που δεν βασίζονται μόνο σε κάποια κριτήρια, αλλά είδαμε πώ μίλησε για διάφορε πτυχέ ο εισηγητή που αφορούν την καθημερινή ζωή όλων των πολιτών. Τώρα, να δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους που είναι συντάκτες δύο θεματικών εγγράφων και θα μας παρουσιάσουν ε, λεπτομερώς τις πτυχές αυτές. Έχουμε τον Αντιπρόεδρο Ταβέρες, ο οποίος θα αναφερθεί ε, στη σχέση της νομιμής παραμονισόδων με τη φοροδιαφυγή και το φορολογικών παραδείσεων. Ο κ. Μπαουργέτσιο θα μας μιλήσει για όλα αυτά που μελετήθηκαν σε σχέση με το ξέπλυμα της τράπεζας και τα χρηματοοικονομικά. Δέκα λεπτά έχετε εσείς, καθώς ε, δεν μακρηγόρησε ο εισηγητής. Ο κύριος Ταβάρες καταρχήν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η κατάσταση που βιώνουμε χαρακτηρίζεται από τρεις μορφές. Καταρχήν ε, έχουμε τεράστιες ανισορροπίες μεταξύ των κρατών της ε, Ένωσης και της Ευρωζώνης και αυτό είναι γνωστό. Δεύτερον, έχουμε τις κυβερνήσεις των χωρών μας, οι περισσότερες από αυτές να βρίσκονται σε αδύναμη δημοσιονομική κατάσταση, σε αδύναμη δημοσιονομική κατάσταση σε επικίνδυνη και κατόπιν έχουμε γενική διάβρωση της εμπιστοσύνης στη δημοκρατία και στους ε, θεσμούς να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή και θα πρέπει να ε, δούμε ότι ο πολίτης αισθάνεται ότι πάντα χάνει και αυτή η αβεβαιότητα οικονομική και θεσμική ε, επιδεινώνεται πολλές ε, φορές γιατί το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βασίζεται πολλές φορές σε νομοποίηση εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και έχουμε συστήσει συστημική φοροδιαφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός ο κύκλος εμποδίζει ε, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, εμποδίζει τις επενδύσεις και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μπορούμε να πούμε ότι τα φαινόμενα αυτά του ξεπλήματος ε, και της ε, φοροδιαφυγής κλέβουν το μέλλον των Ευρωπαίων και οδηγούν στην ανέχεια. Όπως ακούσαμε και τον πρόεδρο Ομπάμα να λέει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ήθελαν να δημιουργήσουν 15 τεχνολογικού τομείς εχμής ε, στις ε, ε, πιο φτωχές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών για να αντιμετωπιστεί κρίση. Λέγαμε ότι θα είναι καλό να κάνουμε το ίδιο και στην Ευρώπη. Ενώ ακούσαμε τον πρόεδρο λέει, να ζητά σύμφωνο ανάπτυξη για την Ευρώπη, το οποίο θα... Ε, έδινε ένα μεγάλο ποσό, αναρωτιόμαστε πού είναι το ποσό, 11 δισεκατομμύρια μίλησε. Πού είναι τα χρήματα λοιπόν, το UNODC, δηλαδή το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για το οργανωμένο έγκλημα και τον μίλησε για το 3% ε, του παγκόσμιου ΕΚΠ ε, χάνεται ε, λόγω της νομοποίησης παρανομενων εισόδων και μιλάμε περίπου για 32 δισεκατομμύρια στο παγκόσμιο ΕΠ. Μόνο στην Ευρώπη αυτό σημαίνει 3% μεταξύ 2 και 3% του Ευρωπαίου ΕΚ και πιστεύουμε ότι το 3 της, ε, σκεφτείτε ότι το 3% είναι το όριο του ελλείμματος ε, για τα κράτη-μέλη μας και ε, χάρη στη φοροδιαφυγή χάνουμε ένα τρισεκατομμύριο της δηλαδή 10 φορές το πακέτο ανάπτυξης του Πρόεδρου Ολάντ. Ο κύριος Γιακολίνο μας έδωσε στο εγγραφό του μία σειρά μηχανισμών μέσω των οποίων γίνεται αυτή η νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων. Έχουμε το καρουσέλ του ΦΠΑ, ε, ψεύτικα τιμολόγια. Επίσης, ε, πολλές φορές παρουσιάζονται ψεύτικα έσοδα από παιχνίδια και διάφοροι μηχανισμοί, διάφοροι είδη μηχανισμών, μεταξύ των οποίων έχουμε και ψεύτικες εταιρείε που ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς ε, σε θηγατρικές ευρωπαϊκών τραπεζών που βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους ε, και κατόπιν ε, μπορούν να ανακτήσουν αυτά τα χρήματα μέσω του ξεπλήματος. Αυτό που πρέπει να επισημαίνουμε είναι ότι οι μηχανισμοί αυτοί χρειάζονται τη συνενοχή του νόμιμου τραπεζικού συστήματος, είτε συνενοχή είτε με παράληψη. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τώρα. Όταν θα αναφέρω τη σειρά των μέτρων που προτείνουμε εμείς στο θεματικό μας έγγραφο για το ξέπλυμα, αυτό ε, σχετίζεται με τη φορολογική εναρμόνιση, με το να θέσουμε τέλος στους φορολογικούς παραδείσους. Εμείς ε, ε θέλουμε να μας πούνε καταρχήν τι κάνουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και πού για να δώσουμε τέλος στους φορολογικούς παραδείσους. ή ε, τράπεζες αν ε, θα μπουν στο μηχανισμό που προβλέπουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ε, πρέπει να μας πούν τι κάνουν οι τράπεζες αυτές και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί τους δίνουμε χρήματα των φορολογουμένων. Δεύτερον, πρέπει να ξέρουμε ποιος έχει τι. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε ένα μητρό σε επίπεδο κρατών μελών που να συντονίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικό και ομοσπονδιακό για τους νόμιμους μετόχους των επιχειρήσεων. Πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις και ποιοι είναι οι μέτοχοι. Και περνάμε εδώ στην τρίτη πρόταση πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι τα άτομα που είναι οι τελικοί δικαιούχοι των περιουσιακών στοιχείων που έχουμε στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες ε, πολλές φορές δεν μας δίνουν τις πληροφορίες. Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό μητρό δηλαδή αυτών των δικαιούχων. Τέταρτον, πρέπει ε, να δούμε ποιος διατάζει. Δηλαδή, όχι μόνο ποιος εργάζεται, αλλά και ποιος διατάζει. Ξέρουμε ότι πολλές φορές είναι ψεύτικες αυτές οι επιχειρήσεις και έχουν κάποιους σκιώδεις ε, διευθυντές, κάποιους σκιώδεις διαχειριστές. Πρέπει λοιπόν ε, αυτοί οι διαχειριστές να λογοδοτούν για τις πρακτικές των δικών τους ε, επιχειρήσεων, αλλά πρέπει να φτάνουμε και στους εντολοδότες. Εμείς ε, βλέπουμε εδώ ότι έχουμε ε, πολλές επιχειρήσεις που πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνες για το τι κάνουν και μάλιστα σε ό,τι αφορά την φοροδιαφυγή, τη φοροαπάτη. Ξέρουμε ότι οι επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν έχουν μεγαλύτερη ισχύ στην αγορά. Επίσης, ε, πρέπει να ενισχύσουμε τη δέουσα επιμέλεια των τραπεζών. Πρέπει να υπάρχει δέουσα επιμέλεια για να ξέρουμε τι απογίνονται τα περιουσιακά στοιχεία που κατατίθεται σε μία τράπεζα. Επίσης, ε, πρέπει να έχουμε και πιο ενισχυσμένη επιμέλεια για τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα. Σκεφτόμαστε πριν τους χάρη τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, κάποιους δικτάτορες αναπτυσσόμενων ε, χωρών. Ε, υπάρχουν ε, τέτοια φαινόμενα. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν την υποχρέωση να ειδοποιούν τις ευρωπαϊκές αρχές όταν υπάρχουν συναλλαγές που υλοποιούνται από τους ανθρώπους αυτούς ε, μέσα στην ενιαία αγορά. Και πρέπει να δίνεται δυνατότητα στις ευρωπαϊκές αρχές ε, να ε, ακυρώνουν αυτές τις συναλλαγές. Αυτή είναι η πρόταση. Και φτάνουμε στην έβδομη πρόταση που αναφέρθηκε ο συγγητής μας σε αυτή. Είναι μια πρόταση την οποία τονίζω να δημιουργήσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, και μέσω της Τραπεζικής Ένωσης σε μια ευρωπαϊκή μονάδα για την έρευνα στο χρηματοοικονομικό τομέα. Αυτή η Ευρωπαϊκή Μονάδα κατά του οικονομικού εγκλήματος θα ερευνούσε όλες τις συναλλαγές ε, πάνω από ένα πασό ή όλες τις ε, διασυνορικές συναλλαγές σύμφωνα με την νομική βάση που υπάρχει στη συνθήκη. Αυτά είναι κάποια μέτρα που θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε. Και για όλα αυτά υπάρχει συνένεση. Δεν αναφέρομαι σε θέματα για τα οποία υπάρχει πολεμική. Και τώρα είναι κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσουμε, γιατί τώρα δημιουργούμε μια τραπεζική ένωση αφενός, αλλά και αφετέρου, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι και μια ένωση δικαίου. Και εμείς ως συνομοθέτες έχουμε τη δυνατότητα να νομοθετήσουμε και στον τομέα του ποινικού δικαίου, της δικαιοσύνης και της ασφάλειας. Επίση, είναι η στιγμή κατάλληλη γιατί μα το ζητάνε οι πολίτε. Αυτή η Δική Επιτροπή έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, λοιπόν, έχοντα ε, κατά νου το αίτημα των πολιτών, αλλά έχοντα και κατά νου τι θεσμικέ εξελίξει. Τώρα έχουμε την αναθεώρηση τη οδηγία για την νομιμοποίηση παράνομων εισόδων, ε, που σύντομα θα περσιστεί Τώρα, τι θα κάνει η Επιτροπή με την οδηγία αυτή, σίγουρα ό,τι κάνει η Επιτροπή θα ληφθεί υπόψη και από τις υπόλοιπες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κυβουλίου ότι είναι Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και την ε, ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, των Ελευθεριών. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Πέρα από την οδηγία που μας παρουσιάζει η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο μπορεί να υποστηρίξει την ερευνητική δημοσιογραφία, που είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να δούμε ποιος ξεπλένει πού βρώμικο χρήμα και πού υπάρχει διαφθορά. Μπορεί να υποστηριχθεί μέσα από πιλωτικά σχέδια που εμείς εγκρίνουμε κάθε μήνα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Μπορούμε να παρουσιάσουμε πιλωτικά σχέδια ως Ειδική Επιτροπή και πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ταμείο για να υποστηρίξουμε την ερευνητική δημοσιογραφία. Επίσης, ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο δούμε ε, τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί, που έχουν δημοφθεί, ε, για να υποστηρίξουμε τέτοια πιλωτικά σχέδια των Ευρωπαίων πολιτών. Η κυρία Μακοβέη παρουσίασε μια πρόταση σχετική, θα άψευστε την Πέμπτη στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και οι ε, συνάδελφοι καλούν να υπάρξει υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας. Τώρα, αυτό που βλέπουμε εμείς είναι η σκοτεινή πλευρά, η εγκληματική πλευρά αυτής της κρίσης και πρέπει να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα αυτά και ως ε, συνομοθέτες ε, πραγματικά μπορούμε να κάνουμε κάτι και πρέπει να το κάνουμε να συμβεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ταβάρες. Και τώρα το λόγο ο κύριος ε, Μποργκέτσο, ο οποίος ε, θα μας μιλήσει για τις σχέσεις παραγωγή παραγωγησόδων με τις τράπεζες. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τις τελευταίες σκέψεις του κυρίου Ταβάρες ε, και των πρότασής του που την υποστηρίζω. Γιατί ασχολούμενος για πρώτη φορά πολύ συγκεκριμένα με το θέμα αυτό που είναι τόσο ευρύ Πρέπει να υπογραμμίσω ότι ο εισηγητής κατάφερε να μας παρουσιάσει ένα εξαντλητικό πλαίσιο μιας θεματικής που πραγματικά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κι άλλη μία πτυχή που πρέπει να υποστηρίξουμε και είναι αυτή που έχει να κάνει με τη δράση του ελέγχου που μπορούν αλλά δεν κατορθώνουν να το κάνουν οι μικροί μέτοχοι όταν συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών ή των τραπεζών, παραδείγματο χάρη. Έχουμε μια πρόσφατη υπόθεση στη δική μας χώρα και ακόμη και ένα τυφλός θα καταλάβαινε πως ε, πολλές φορές ε, οι μικροί μέτοχοι δεν μπορούν να ασκήσουν τέτοιες δραστηριότητες ε, ελέγχου. Επομένως, θα πρέπει να κατορθώσουμε να κάνουμε να λειτουργήσει ένα σύστημα το οποίο από νομική σκοπιά φαίνεται ήδη πολύ προχωρημένο, πολύ προηγμένο. Αν εμεί δούμε όλη τη διαδρομή από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι σήμερα, έχουμε σημειώσει πρόοδο, είχαμε συμβάσει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τώρα περιμένουμε μία νέα οδηγία που θα περιλαμβάνει τις νέες συστάσεις της ΓΚΑΦΗ, της Task και επίσης με τις συστάσεις της ΓΚΑΦΗ και τις επικαιροποίησεις ε, θα έλεγα ότι μιλάμε για μία συνεχή εξέλιξη της ε, επιδεξιότητας και το λέω με αρνητικό τρόπο του ε, οργανωμένου εγκλήματος ε, και των τρομοκρατικών ομάδων που χρησιμοποιούν το εργαλείο του ξεπλήματος. Τίθεται όμως ένα ερώτημα. Γιατί έχουμε τόσο, τόσο λίγα αποτελέσματα παρά το νομικό πλαίσιο. Πρέπει εδώ να αναλύσουμε το κενό που υπάρχει μεταξύ των, διάφορων πτυχών του φαινομένου το UNODC το 2009 μας μιλάει για 2 δισεκατομμύρια δολάρια που κατασχέθηκαν και επίσης Έχουμε και το σκάνδαλο της HSBC στις Ηνωμένε Πολιτείε που έφτασε σε ένα πρόστιμο 1,9 ε, δισεκατομμύρια δολάρια και ε, για την έρευνα της Bank of America, της Τράπεζας ε, της Αμερικής και επίσης έχουμε και άλλες έρευνες που αφορούν τη UBS και την Deutsche Bank στη Φραγκφούρτη. Εγώ πιστεύω λοιπόν, εξετάζοντα ε, μόνο αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία, κατανοούμε πόσο πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα ε, στη φαινομολογία της νομοποίησης παράνομων εσόδων. Στη σύνοδο του ΙΕ ε, για την ε, παγκόσμια διακίνηση σε ναρκωτικών ουσιών. Εκεί και ότι δεν θα ήταν ε, δυνατό να έχουμε διεθνείς συναλλαγές των μεγάλων εμπόρων ναρκωτικών χωρίς οι τράπεζες να διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Και από αυτή τη σκοπιά φαίνεται προφανές ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε συγκεκριμένα εργαλεία για την καταπολέμηση. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι πάντα εκ των υστέρων υπάρχει παρέμβαση. Και αν βλέπουμε μια τόσο μεγάλη τράπεζα όπως η HSBC να αναγκάζεται να πληρώνει ένα πρόστιμο 1,9 δισεκατομμύρια, μπορείτε να φανταστείτε τι έχει γίνει στο παρελθόν. και τα στοιχεία σε σχέση με το οικονομικό όφελος Δηλαδή, στις περιπτώσεις που έχει μελετηθεί όλη η δραστηριότητα της Κόζα Νόστρα και άλλων, βρίσκουμε ότι καλύπτονται όλα τα στοιχεία, ότι υπάρχει ομερτά, υπάρχει συγκάλυψη, υπάρχει αδυναμία να σκάψουμε εις βάθος. Και υπάρχει προστασία ουσιαστικά του τραπεζικού συστήματος. Έτσι λοιπόν η δική μας ε, προσέγγιση θα πρέπει να επικεντρωθεί και στην ανάλυση των λαθών που έχουν γίνει και των κενών που επιτρέπει η νομοθεσία. Πρόκειται για μια προσέγγιση που δεν αιτιολογείται πάντα από το τραπεζικό σύστημα, ε, παραπονιέται για κόστος. Για το κόστος που επιφέρουν ε, οι δραστηριότητες ελέγχου. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει οι ελεγκτικές δράσεις και καταγγελίας να γίνουν πιο αποτελεσματικές και πιο ταχύς δεν ε, μας εξυπηρετεί το να έχουμε χιλιάδες κανόνες που προκαλούν σύγχυση. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι συγκεκριμένα πρέπει να στοχεύσουμε εκεί όπου χρειάζεται και να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε εκεί όπου χρειάζεται. Και ο κύριος Σταβάρες πολύ σωστά μας ανέφερε διάφορες περιπτώσεις, την περίπτωση των ε, PEPs, των πολιτικών προσώπων που εκτίθενται, αλλά θα πρέπει και να επικεντρωθούμε, το χάρη, και σε συναλλαγές ε, όπου ενέχονται άνθρωποι που προέρχονται από τρίτες χώρες. βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά πρόσωπα από τις χώρες αυτές, ε, κάποιοι δικτάτορες, παραδείγματος χάρη αφρικανικών χωρών, και μπορεί να συμμετέχουν ακόμη και σε παγκόσμιες μασονικές οργανώσεις. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε εκεί περισσότερο, να δούμε τι κάνουν αυτοί, παρά να επικεντρωθούμε ε, σε κάποιον ε, μικροεγκληματία που μπορεί να δραστηριοποιείται στο Παιδεμόντιο, παραδείγματος χάρη. και που μπορεί να προβαίνει σε φοροδιαφυγή. Αυτή είναι η προσέγγιση που η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα πρέπει να ξεκινήσει να έχει και κατά την ταπεινή μου γνώμη μέχρι τώρα δεν ήταν ορθή η προσέγγιση, δεν είχε τα κατάλληλα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη ικανοποιητικά. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει και άλλη μια σημαντική πτωχή που πρέπει να μας καθορίσει, δηλαδή το πώς σχετίζεται αυτή η δραστηριότητα της δρομοποίησης παράνομων εσόδων με την άρση, ε, την κατάργηση της ισορροπίας των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Βλέπουμε ε, ποσά που είναι ανεξέλεγκτα, που προέρχονται από παράνομες πηγές και μέσω της, ε, του ξεπλήματος μπαίνουν στην νόμιμη οικονομία και όλο αυτό σημαίνει αθέμητο ανταγωνισμό. Και ο αθέμητος ανταγωνισμός βλάπτει το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματιών που δεν έχουν ε, τέτοιες ε, δυνατότητες ε, και μάλιστα σε περιόδους τέτοιας οικονομικής κρίσης δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τις τρόπεζες με χαμηλά επιτόκια. Επομένως, ε, είναι πολύ σημαντικό για όλους ε, όσους ε, θέλουν να λειτουργεί η οικονομία βάσει ενός υγιού συστήματος μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που παράγουν και δημιουργούν θέσεις εργασίας να προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε όλες αυτές τις παράνομες δραστηριότητες. Έχουμε και κάποιες ενδείξεις, ε, κάποιες προτάσεις της ΓΚΑΦΗ που πρέπει να μεταφραστούν σε συγκεκριμένα μέτρα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε και τις φωνές από τον τραπεζικό τομέα. Στη χώρα μας είχαμε μία φωνή πολύ θετική, γιατί και από τον τραπεζικό κόσμο εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα θετικό και υγιές κύκλωμα που είναι το ε, ευρωπαϊκό σύστημα των λαϊκών τραπεζών, των συνεταιριστικών τραπεζών. Σε τέτοια κυκλώματα πολλές φορές βλέπουμε να υπάρχουν τέτοιες ε, ύποπτες συναλλαγές, ακόμη και εκεί, αλλά αυτές τις δραστηριότητες συνήθως ε, χαρακτηρίζουν τις τράπεζες που κερδοσκοπούν και αν ε, δεν ε, διαχωρίσουμε αυστηρά ε, σύμφωνα με το δόγμα του Ρούσβελτ, τις τράπεζες, τις εμπορικές από τις παραδοσιακές τράπεζες, τότε θα συνεχίσει το φαινόμενο αυτό και δεν θα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όποια νομοθεσία και αν επινοήσουμε. Αυτή είναι μια κύρια αρχή, μια βασική αρχή εμείς ε, θέλουμε να θεραπεύσουμε το κακό, αλλά αυτό εξαρτάται από αυτή την πολύ σοβαρή στρέβλωση που είναι μπροστά στα μάτια μας. Και δεν βλέπουμε να υπάρχει συγκεκριμένη βούληση από τις ευρωπαϊκές αρχές ε, να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις. Προφανώς ε, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα Μπορούμε να δούμε κάποιες ε, περιπτώσεις, ε, παραδείγματος χάρη, ε, στα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια έχουμε ένα μακροσκοπικό φαινόμενο. Δηλαδή, διάφορες εγκληματικές οργανώσεις κάθε είδου εκμεταλλεύονται κάποια κενά που υπάρχουν και κάποιες καινοτομίε που δίνονται βάσει του εξυγχρονισμού των συστημάτων στο διαδίκτυο. Και ε, οι διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο αυτό θα πρέπει να ανοίξει τα μάτια ε, στους νομοθέτες που καθυστερούν πάρα πολύ ακόμη. Γιατί έχουμε εκεί ένα τεράστιο χώρο φοροδιαφυγής. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Μποργκέτσιο. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια σύνθεση των παρεμβάσεων ε, των συναδελφών Ταβάρες και Μπορκέτσιο. Δηλαδή υπάρχει ένας κοινό παρανομαστής, η αναγκαιότητα διαφάνειας. Και αυτό μας ε, οδηγεί είτε στη διαφάνεια των μικρών συναλλαγών, είτε στο να ξέρουμε την πραγματική ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων. Διαφάνεια σε σχέση με τις επιχειρήσεις ε, και μεγάλων και μικρών. Γιατί δεν έχουμε μόνο το πρόβλημα με τις πολυεθνικές, ε, αλλά και κάποιων μικρών επιχειρήσεων έχουμε ένα φαινόμενο μπάμπουσκας. Πολλές ε, φορές ε, αστυνομικές επιχειρήσεις μας έχουν δείξει ότι υπάρχει το φαινόμενο αυτό. Τώρα να ξεκινήσω τη συζήτηση, να δώσουμε το λόγο στους συντονιστές. Για το ΕΛΚ, Ματιέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τους εισηγητές τον κύριο Γιακολίνο με την επόμενη του, με την τελευταία του θεματική έκθεση που ακολουθεί τις τρεις προηγούμενες. Καθώς και για τις προτάσεις που μας έκανε για το σημερινό θέμα το ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος και την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων. Στην έκθεση αυτή λοιπόν γίνεται, δίνεται ένας ορισμός και αυτό είναι σημαντικό γιατί και οι εμπειρογνώμονες έχουν πρόβλημα να καθορίσουν τη σωστή, το σωστό νομικό υπόβαθρο και οι ορισμοί που μας δίνει σήμερα ο εισηγητής είναι πολύ χρήσιμοι. Οι προτάσεις του, οι συστάσεις του με βρίσκουν σύμφωνοι, ιδιαίτερα η προσοχή που δίνει στις ε, διαμεθοριακές μεταφορές ως προς το ξέπλυμα, καθώς και τους φορολογικούς παραδείσους και την τραπεζική λεγόμενη διακυβέρνηση. Η φορολογική, δημοσιονομική εναρμόνιση είναι κάτι που πρέπει να το προτείνουμε και στο Συμβούλιο γιατί εκείνο τώρα πρέπει να αντιδράσει. Πρέπει λοιπόν να το πράξει. Ο Νικόλαος Σαρκοζή, αν θυμάμαι καλά, το 2008, είχε ήδη τονίσει στην Ένωση και το είπε και ο κύριος Σταμπάρες νομίζω ότι δεν έχει περάσει ακόμα η κρίση ως προς τους φορολογικούς παραδείσους και από τότε που τα είπε ο Σαρκοζή τίποτα δεν έγινε. Πρέπει λοιπόν ίσως να σκληρύνουμε κάπως τη στάση μας στην έκθεση αυτή για να πιστεί πιο εύκολα το Συμβούλιο. Άλλη σύσταση που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε είναι σε συμφωνία με τους δικηγόρους και με τους δικηγορικούς συλλόγους να κάνουμε κάτι γιατί είναι εκπληκτικό ότι η μαφία στηρίζεται από ορισμένους φορολογικούς δικηγόρους που δεν ακολουθούν φυσικά καμία από την θεμητές δεοντολογίες που είναι γνωστές και υποφελούνται από την νομοθεσία που ισχύει για την προφυλάκηση κλπ. Βέβαια, πολύ σεβαστή, σεβαστό επάγγελμα είναι εκείνο του δικηγόρου, αλλά ως προς το ξέπλυμα του βρωμίκου χρήματος θα έπρεπε νομίζω να ξεπληθεί λίγο και το επάγγελμα αυτό και να το λέμε στην εκθέσή μας θα ήθελα. ως προς την ανεύθυνη συμπεριφορά ορισμένων τραπεζών και αυτό πρέπει να το πούμε, συμφωνώ και επειδή μίλησε γι' αυτό και ο κύριος Ταβάρες σε ορισμένες χώρες δικτατορικές υπάρχουν προβλήματα ως προς την απορρόφηση και χρησιμοποίηση των ενωσιακών κονδυλίων. Θυμάμαι ότι είχα πάει στο Αφγανιστάν κάποτε με την Κοκομπού για να δω ποια είναι η χρήση, να δούμε ποια είναι η χρήση των ενωσιακών κονδυλίων και διαπιστώσαμε ότι τα μετέφερε εκεί η Παγκόσμια Τράπεζα, τα διαπίστωνε, τα επαλήθευε η Κομισιόν τοπικά και κατέληξε η Κοκομπού ότι δεν υπάρχει καμία παραβίαση ούτε παρατυπία. Ενώ διαπιστώσαμε ότι τελικά υπάρχει κατάχρηση, κακή χρήση των ενωσιακών κοντιλίων και η Εύα Ζολή που είχε πάει τελευταία εκεί διαπίστωσε και εκείνη ότι παρά τις προσπάθειες της Κομισιόν και της Παγκόσμιας Τράπεζας γίνεται και εκεί ξέπλυμα βρωμίκου ευρωπαϊκού χρήματος. Ενώ βέβαια από τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Κομισιόν φαίνονταν όλα σωστά και ότι όλα διατίθενταν εκεί όπου έπρεπε. Σας ευχαριστώ και αναμένω τα υπόλοιπα σχόλια και μπράβο για τη δουλειά σας. Ευχαριστώ κυρία Ματία. Δεν ξέρω ο κύριος Νιτοντάν, θέλει το λόγο. Um, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που κάνετε τόσο μεγάλο έργο για να γράψετε το σχέδιο αυτό της έκθεσης. Είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες και πολύ χρήσιμες, μεγάλη πηγή ε, χρήσιμων πληροφοριών. Σας συγχαίρω. Νομίζω ότι το θέμα αυτό αποτελεί την καρδιά, αν θέλετε, και τον πυρήνα των προβλημάτων. Γιατί τα χρήματα τα οποία χάνουμε με όλους αυτούς τους τρόπους. Στο παράρτημα 1 έχουμε ένα πολύ χρήσιμο κατάλογο για το πώς μπορεί να γίνει νομιμοποίηση εσόδων. Σας ευχαριστώ. Σελίδες ολόκληρες για ξέπλυμα χρήματος. Όλα αυτά λοιπόν καταστρέφουν θέσεις εργασίας, ε, νόμιμα έσοδα για τα κράτη-μέλη και για την Ένωση. Αν λοιπόν δεν μπορούμε να τα ανακτήσουμε τα χρήματα αυτά, θα ε, τα χάσουμε, θα αιμορραγήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να περάσουμε και πέρα από την, ε, το ξέπλυμα του χρήματος που είναι ε, παράνομο, να συμπεριληφθούν και η φορολογική παράδειση που είναι νόμιμη. Γιατί όσο υπάρχουν και είναι νόμιμοι, ακόμα και αν λάβουμε άλλα μέτρα, τα χρήματα αυτά μπορούν να πάνε στα νησιά και οι σε οποιοδήποτε άλλο φορολογικό παράδεισο. Άρα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα μπροστά μας. Τρία πράγματα λοιπόν έχω γράψει, τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να μπουν στην έκθεση. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα πετύχουμε, γιατί έχουμε και την κοινή γνώμη. Αν η Επιτροπή μας καταφέρει να κερδίσει την κοινή γνώμη την ευρωπαϊκή, θα καταφέρουμε πολλά, γιατί θα οθήσει έτσι η κοινή γνώμη τις κυβερνήσεις του να αναλάβουν μέτρα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν κεντρικές αρμοδιότητες στις Βρυξέλλες, γιατί μπορεί τα 27 κράτη-μέλη να είναι σε θέση να έχουν νομοθεσία, δράσεις, ξεχωριστές, αλλά η χώρα που γνωρίζω εγώ καλύτερα από είναι η καλύτερη στο ξέπλυμα χρήματος. Χρειαζόμαστε λοιπόν από τις Βρυξέλλες να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο ισότιμου ανταγωνισμού, αν θέλετε και θεωρώ, Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και να αντιγράψουμε αυτά που εφαρμόζονται στη ΣΥΠΑ για τα extraterritoriality, για την εξωτερική διάσταση της ε, σε ό,τι αφορά την ετεροδικία για τους Ευρωπαίους πολίτες εκτός των ευρωπαϊκών ε, συνόρων. Και αν το καταφέρουμε αυτό, νομίζω ότι θα κάνουμε μεγάλο βήμα στο και μεγάλη πρόοδο. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι τα έγγραφα αυτά αποτελούν μια πάρα πολύ καλή βάση και μια πάρα πολύ καλή πηγή πληροφοριών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντοντάν. Παρακαλώ, κύριε Καρόνα. Ένα λεπτό μόνο για να εκφράσω δύο σκέψεις. Καταρχήν να πω πόσο εκτιμώ το έργο των συναδέλφων και επίσης ε, να πω πως σκεφτεί ότι υπάρχει μεγάλη συμφωνία για αυτό το έργο. Υπάρχει λοιπόν μια καλή βάση για να αναλάβουμε δράση. Δεύτερον, σε σχέση με όσα είπε η κυρία Ματιέ, πιστεύω, αλλά ίσως αυτό να το σκεφτούν οι συγητές καλύτερα, ίσως θα ήταν σκόπιμο να υπογραμμίσουμε περισσότερο την αναγκαιότητα δέσμευσης μιας προσοχής που πρέπει να δοθεί, μιας επαγρύπνησης. Θα το βρούμε τέλος πάντων τον όρο από την πλευρά των δικηγόρων, από ε, τις ε, εμπορικές ενώσεις, τους συλλόγους τους εμπορικούς, γιατί, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Ιταλία, σε κάποιες περιοχές ε, στη Βόρεια Ιταλία οι άνθρωποι αυτοί διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι αυτοί οι σύλλογοι πρέπει να διαδραματίσουν πιο αποφασιστικό ρόλο σε σχέση με το ρόλο που έχουν διαδραματίσει μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε κύριε Καρόνα, ναι και εγώ θεωρώ να βασιστούμε στην πρόταση της Βερονίκ αυτό είναι κάτι που είναι ενώπιόν μας και δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για την Ιταλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο οι κατηγορίες αυτές έχουν διδραματίσει σημαντικό ρόλο για τις δραστηριότητες του οργανωμένου κλίματος και στο μακρινό Λονδίνο αν θέλετε που είναι μακριά από ε, το επίκεντρο και εκεί έχουμε ε, πολύ δραστηριότητες σε τέτοιο βαθμό και διαδραματίσουμε πώς ε, ε, διαδραματίσουν ένα όλο ένα και μεγαλύτερο ρόλο οι δημόσιοι ε, υπάλληλοι αλλά και η δικαστική αρχή, η ερευνητική αρχή θα πρέπει να βλέπουν που παρέχονται κάποιες υποσχέσεις, ε, κάποιες, ε, κάποια ανταλλάγματα. Έτσι λοιπόν, αν είναι δυνατόν ε, και στην έκθεση της Επιτροπής αυτής, στην έκθεση του κυρίου Γιακολίνου, να προσπαθήσουμε να δείξουμε πόσο αδιάλακτοι είμαστε έναντι των ευθυνών που έχουν άλλοι και να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια μήνυματα άλλης φύσης. Σε σχέση με αυτό που θα θέλαμε εμείς από μια τόσο σημαντική κατηγορία. Υπάρχει και άλλη μια πτυχή. Εμείς πολλάκις το συζητήσαμε αυτό το θέμα στην Επιτροπή αυτή και εγώ θα επαναλαμβάνω ότι αυτή η Επιτροπή μέχρι σήμερα έχει κάνει μια αξιοσημείωτη δουλειά γιατί εμβάθυνε σε όλα τα θέματα που για τόσα χρόνια στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ δεν ήταν δυνατόν να εμβαθύνουν επειδή δεν υπήρχε χρόνος. Όμως εμείς ε, μιλήσαμε για συγκεκριμένα θέματα και προλίγου εισηγητής, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ο κύριο Σταβάρες ίσω νομίζω, είπε ότι την Πέμπτη το πρωί εμείς θα ψηφίσουμε στη Λίμπε την έκθεση της κυρίας Μακοβέη για την οδηγία περιδίμευση. Πόσες φορές στη Λίμπη μπορέσαμε να μιλήσουμε για το περιεχόμενο, για την αναγκαιότητα και πόσες φορές ε, στο ιστορικό αυτής της επιτροπιστικής μας εκράσεις μιλήσαμε για τα θέματα αυτά. Εμείς πραγματικά λεπτομερώς εξετάσαμε όλα όσα μπορούσαν να μας πούν εμπειρογνώμονες για τη δίμευση, για την κατάσχεση, για τη χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων για κοινωνικούς σκοπούς. Και αυτό είναι σημαντική πτυχή της δίμευσης και της κατάσχεσης. Αν ε, αυτό το κοινοβούλιο δεν έδινε την πρέπουσα αξία στη χρήση των περιουσιακών στοιχείων για κοινωνικούς σκοπούς θα κάναμε τεράστιο λάθος. Επομένως, αυτή η Επιτροπή έχει κάνει ό,τι μπορούσε να κάνει. Ε, συζητήσαμε θέματα που ήταν σχεδόν άγνωστα και πραγματικά ασχοληθήκαμε με γιατί το μοναδικό μας ε, ε, ενδιαφέρον είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε τα κατάλληλα εργαλεία, τα κατάλληλα μέσα για να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα. Ο ρόλος των τραπεζών και ο ρόλος των φορολογικών παραδείσων. Ακόμη και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν μαύρες τρύπες. Υπάρχουν ε, κάποιες καταστάσεις που όχι μόνο θα πρέπει να μας προβληματίζουν και να μας προκαλούν ντροπή, γιατί από δημοκρατική σκοπιά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε χρηματοοικονομικά σκάνδαλα όπου εμπλέκονται φορολογική παράδεση εντός ε, της δικής μας επικράτειας και δεν μπορούμε να πάμε μακριά ε, αρκεί να θυμηθούμε κάποια σκάνδαλα δεν μπορούμε να ξεχνάμε το ρόλο του Λουξεμβούργου και της Ελβετίας η Ελβετία δεν αποτελεί μέρος της Ένωσης, έχει όμως ένα θεμελιώδη ρόλο. Λίγο καιρό πριν αποφάσισε να είναι κάπως πιο σαφής, πιο ξεκάθαρη, να προσφέρει κάπως ε, περισσότερα στοιχεία που να διευκολύνουν τις ερευνητικέ αρχές, όμως είμαστε ακόμη μακριά από τους στόχους που έχουν τεθεί. Είναι απαραίτητο και κρίσιμο όχι μόνο να έχουμε μια διαφάνεια ε, έναντι κάθε χρηματοοικονομικής συναλλαγής ε, όπως είπε και η κυρία Ματιέ, αλλά να υπάρχει και διαφάνεια στο πώς χρησιμοποιούνται οι ευρωπαϊκοί πόροι. Και αυτή την τυχή την έχουμε συζητήσει πολλάκις, αλλά αφορά πάρα πολύ και τη δική μας οικονομία, τους δικούς μας πόρους. Και πολύ συχνά εγώ όταν ε, βλέπω κάποιες ανομοιογένειες πραγματικά τα χάνω. Στην Σικελία υπάρχει ένα επίπεδο ε, πολύ χαμηλό για προειδοποίηση που Πότε ε, γίνεται αυτή η προειδοποίηση, όταν έχουμε κάποιες περιοχές όπως η Κελία, Καλαβρία, περιοχές του στόχου 1, υπάρχουν ε, αυτοί οι συναγερμοί, ακόμη και αν υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες από τις ε, ερευνητικές αρχές. Επομένως, Όταν ε, μιλάμε για τους σπόρους που παρέχονται σε αυτές τις περιοχές, ε, μιλάμε για σημαντικά ποσά και γίνεται συνέχεια αξιολόγηση από το ελεκτικό συνέδριο, από τις ε, διάφορες δικαστικές και ερευνητικές αρχές. Όμως με εκπλήσει το γεγονός με εξέπληξε το γεγονό ότι στην Γερμανία αυτό το επίπεδο είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Δηλαδή ο συνεγερμός ε, εμφανίζεται μετά όταν έχει εξαφανιστεί το ποσό. Και μήπως αυτό θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε, δεν θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε ότι δεν υπάρχει υπεξαίρεση στη Γερμανία επειδή δεν υπάρχει ο έλεγχος, αλλά ο έλεγχος αυτός θα έπρεπε να είναι ομοιόμορφος, όλοι θα έπρεπε να έχουμε την ίδια θέση όταν ε, ουσιαστικά υπάρχουν υποψίες ε, για κακοδιαχείριση ή υπεξαίρεση χρήματος. Στο παρελθόν ε, είχαμε μία μη δυναμική θέση, όμως εδώ έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε και σε σχέση με τις νέες χώρες που θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε και να αξιολογούμε μία σειρά καταστάσεων που θα παρουσιαστούν με την προσχώρηση των νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μία πρόκληση. Δεν μπορούμε να είμαστε προετοίμαστοι ενώπιον αυτής. Και μάλιστα αυτή η Επιτροπή την έχει κατανοήσει από την αρχή και το να έχει κατανοήσει κανείς μία τόσο σημαντική πρόκληση να σας υπενθυμίσω ότι στην πρώτη ακρόαση εμπειρογνώμονες που κάθισαν σε αυτό το τραπέζι τόνιζαν πόσο σημαντικό είναι και φαινόταν ε, και σαν να παρουσιαζόταν ένα στόπ τότε το πόσο πολύπλοκα είναι τα διάφορα νομικά συστήματα αυτή πρέπει να είναι λοιπόν η σημαντική πτυχή, το σημαντικό, πιο σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης που θα μας κάνει να κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια σοβαρή Ευρωπαϊκή Ένωση αν ε, δεν ε, ενοποιήσουμε τα συστήματα που είναι τόσο πολύ σημαντικά για τη συμβίωση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πέρα από τις δημοκρατικές αξίες μιλώ για τα στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια και μάλιστα την χρηματοοικονομική και την οικονομική ασφάλεια. Στην οικονομία μας πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν μπορεί να δεχτεί από κανέναν επίθεση. Ούτε θα μεταμορφωθεί από νόμιμη σε παράνομη οικονομία. ούτε πρέπει να κάνουμε αυτή την παράνομη οικονομία θεσμό. Τώρα, θα δώσω το λόγο στους εισηγητές για να απαντήσουν στις παρατηρήσεις. Παρακαλώ, κύριος Γιακολίνο. Άκουσα την παρέμβαση όλων ε, όσων ε, συνέσφεραν και του κυρίου Ταβάρης, του κυρίου Μποργέτζου. σε πάρα πολλές πτυχές. Υπάρχει συμφωνία απόλυτη για τις δραστηριότητες. Άκουσα βέβαια και τις παρεμβάσεις της κυρίας Ματιέ και τις προτάσεις της για την συνεργασία, για την προσφυγή στη βοήθεια ορισμένων επαγγελματικών κατηγοριών. Άκουσα και τους κυρίους Καρουνό και Νιτοντάν. Είμαστε στο σωστό δρόμο για να έχουμε ένα κείμενο που μπορεί να αντικατοπτρίζει τις ε, προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Μάλιστα. Ο κύριος Ταβάρης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους ε, αυτές τις συγκεκριμένε ερωτήσεις για το θέμα των δικηγόρων. Για το θέμα των δικηγόρων, στους οποίους αναφέρθηκε η κυρία Ματιέ είτε μιλάμε για μεμονωμένους ε, πολίτες που φοροδιαφεύγουν, είτε για εγκληματικέ οργανώσεις που φοροδιαφεύγουν, ε, πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους φορολογικούς παραδείσους και αυτούς που υπάρχουν μάλιστα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πολύ μεγάλο μέρος ε, της φοροδιαφυγής ε, γίνεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιούνται διάφορες εθνικές δικαιοδοσίες ή χρησιμοποιείται το ότι υπάρχει ε, διαφορετική κουλτούρα τραπεζική μεταξύ των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να ξέρει και η γνώμη και οι είναι ότι τελικά τι γίνεται μέσω αυτών των διαδικασιών, ότι υπάρχουν φόροι πιο υψηλοί για όλους. Γιατί αν ε, δεν ε, κατορθώσουμε να αφαιρέσουμε το οξυγόνο από τις πρακτικές αυτές, εμείς ε, μπορούμε να αφαιρέσουμε το οξυγόνο με πολλές φορές. Γιατί, ε, το οξυγόνο αυτών είναι η αδιαφάνεια στη χώρα μου, παραδείγματος χάρη, ε, να έχουμε μία συγμένη υπηρεσία ε, συγγνώμη, μια εισηγμένη τέτοια περίπτωση υποχρεούται να δίνει πληροφορίε ε, αυτή η επιχείρηση. Ενώ στην Ολλανδία δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εμεί πρέπει να λέμε τώρα ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δινει πληροφοριε αυτη η επιχειρηση ενω στην ολλανδια δεν συμβαινει κατι τετοιο εμει πρεπει να λεμε τωρα οτι σε ολη την ευρωπαικη ενωση πρεπει να ισχυει το ίδιο καθεστώς για τις επιχειρήσεις για να προστατεύουμε τον καταναλωτή και τον πολίτη. Όμως ε, το δικό μας ε, φορολογικό σύστημα ε, δεν μπορεί τελικά να καταλήξει σε μικρότερη φορολογία για τους πολίτες αν δεν το αντιμετωπίσουμε αυτά, ούτε μπορούμε να έχουμε επενδύσεις. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι πρέπει αυτό το θέμα να το δούμε από ποια σκοπιά και αν το δούμε, είτε προοδευτική είτε συντηρητική, από μία νομική σκοπιά δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι προσφεύγουν στον νόμιμο τομέα της οικονομίας μας, στις τράπεζες δηλαδή, και, στην, ε, και στους δικηγόρους για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν κατόπιν κανάλια που χρησιμοποιεί το ίδιο το οργανωμένο έγκλημα, όπως ε, το χάρη άνθρωποι που προβαίνουν σε εμπόριο ναρκωτικών, ε, εμπόριο ανθρώπων, εμπόριο όπλων. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει όλοι αυτοί οι πόροι να διοχετευτούν στο νόμιμο τμήμα της οικονομίας. Και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι ε, σημαντικό να διερευνηθούν τα δικήματα αυτά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίσης, ε, η απάτη με τους κοινοτικούς πόρους Πρέπει να διερευνηθεί το θέμα αυτό, γιατί πολλέ φορέ ακούσαμε ότι υπάρχει παράνομη χρηματοδότηση των κομμάτων, χρησιμοποιούνται εκεί πόροι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του κοινοτικού προπολογισμού. Και θα πρέπει λοιπόν αυτό να καταστεί αδίκημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση τώρα με τα θέματα που έθεσε ο κ. Νιούτον Ντάν. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να κερδίσουμε την κοινή γνώμη. Νομίζω ότι ε, πρέπει η κοινή γνώμη να κερδίσει εμάς. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται και στο Συμβούλιο, όπου δεν εκλέγονται εκεί οι πρόσωποι. Επομένως, πρέπει τελικά να εξυπηρετήσουμε το ευρωπαϊκό συμφέρον. Και τέλος η χώρα μου, η Πορτογαλία, χάνει 2 δισεκατομμύρια λόγω της φοροδιαφυγής, της φοροαπάτης ετησίως. Και όλα τα έσοδα από τη φορολογία είναι 15 δισεκατομμύρια. Δηλαδή χρειαζόμαστε ε, τρία χρόνια για να ανακτήσουμε όλα όσα χάνουμε μέσα σε ένα χρόνο. Και ξέρετε ότι δεν αναπτυσσόμαστε όλας. Αυτά τα φαινόμενα, αν δεν τα λύσουμε τώρα, αυξάνουμε το μέγεθος της επόμενης χρώσης που αναπόφευκτα θα έρθει. Ευχαριστώ Ρούι. Και εγώ συμφωνώ ότι αυτές είναι αιτίες της κρίσης, όχι το αποτέλεσμα. Ο κύριος Μπορκέτσι. Ευχαριστώ. Οι παρατηρήσεις που ακούστηκαν συγκλίνουν όλες. σε στόχους που έχουν χαρακτηρίσει το έργο αυτής της Επιτροπής. Φυσικά συμφωνώ με το πνεύμα και με την ποιότητα των συμπερασμάτων που υπάρχουν στο έγγραφο του εισηγητή. Και θα ήθελα και να υπενθυμίσω και το πόσο οι υπηρεσίες μας βοήθησαν και στο συντονισμό αλλά και στην ενημέρωση. Παραμένει σε μένα πεποίθηση ότι πέρα από την ε, περαιτέρω εκπόνηση των νομικών μέσων πρέπει να μιλήσουμε και για την πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά το φαινόμενο πέραν ε, των διαφόρων ιδεολογιών. Γιατί εδώ ενέχονται πάρα πολύ σοβαροί κίνδυνοι για την νόμιμη οικονομία μας. Και είδαμε και ποιες είναι οι συνέπειες. Μιλήσαμε για την περίπτωση της Πορτογαλίας, για την ε, φοροδιαφυγή. Όμως ε, έχουμε συνέπειες σε πάρα πολλούς τομείς. Και καθώς τώρα είμαστε σε εκλογική περίοδο στην Ιταλία, δεν θέλω να κατονομάσω, όμως οι Ιταλοί συνάδελφοι γνωρίζουν πολύ καλά το τι συμβαίνει και έχουμε και τις περιπτώσεις που μας δείχνουν ότι ο κύριος οργανισμός εθνικού ελέγχου, δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα μιας χώρας, δεν αντιλαμβάνεται ότι σε μία από τις κύριες χώρες της ίδιας χώρας είχαμε συναλλαγές ε, εκατομμυρίων ευρώ που δεν ήταν καθόλου νόμιμες ούτε διαφανείς για τα παράγωγα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, ε, υπάρχει μεγαλύτερο σύνδεσμος και με τη διαφθορά και όχι τόσο με το οργανωμένο έγκλημα, σε αυτή την περίπτωση, ευτυχώς. Αλλά τίποτα δεν μας κάνει να σκεφτόμαστε Ενώ εμεί μιλάμε ότι δεν υπάρχουν τέτοια χειρότερα φαινόμενα έτσι. Λοιπόν, αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να μην λειτουργεί αυτό το σύστημα. Και πώς είναι δυνατόν οι ίδιοι οι ελεγκτικοί οργανισμοί να μην υλοποιούν αυτό που πρέπει να κάνουν. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει εμείς ε, να εφεύρουμε κάποια μέσα που να μας ε, επιτρέψουν να αποφύγουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν σημαίνει ότι ό,τι λειτουργεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι καλύτερο από αυτό που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο. Μπορεί και τα δύο να πηγαίνουν σε λανθασμένη κατεύθυνση. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε την ε, εμπειρία και των πολύ σοβαρών ε, παραλήψ, για τις πολύ σοβαρές παραλήψεις και λάθη που έχουμε σε εθνικό επίπεδο και ε, που δυστυχώς πολλαπλασιάστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, αν έχουμε σε μια κεντρική τράπεζα τέτοιες παραλήψεις, τότε ε, κατανοείτε ποιες είναι οι συνέπειες ε, των όσο δεν κάνουν οι κυβερνήτες των τραπεζών. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νιούτον Σύντομα, σύντομα. Ήθελα να πω στον φίλο μου τον Αντιπρόεδρο Ταβάρες που είπε ότι δεν χρειάζεται καμία καμπάνια για την κοινή γνώμη, αν κατάλαβα καλά, γιατί είπε ότι ο κόσμος γνωρίζει ήδη τα πράγματα, διαφωνώ. Νομίζω ότι η κοινή γνώμη τοπικά μπορεί να ξέρει εκεί όπου ζει ο καθένας, αλλά δεν έχει καμία γνώση του, της κλίμακας για την οποία συζητάμε εδώ. Και αυτό πρέπει να τους πούμε, γι' αυτό πρέπει να τους πληροφορήσουμε, ότι όλα αυτά είναι πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων από ό,τι νομίζαμε στο χωριό μας ή στη χώρα μας οι εθνικές κυβερνήσεις δεν είναι διατεθειμένες να κάνουν κάτι, να αναλάβουν μέτρα για να διορθώσουν τα πράγματα παρά μόνο όταν πιεστούν, παραδείγματος χάρη, για το κρέας αλόγου που ξαφνικά έχει γίνει το πιο ενδιαφέρον θέμα στην Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις λένε όλες κάτι θα πάρουμε μέτρα, αυτό το κάνουν επειδή δόθηκε δημοσιότητα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει αν θέλουμε οι εθνικές κυβερνήσεις να κάνουν κάτι, να αντιδράσουν για το οργανωμένο έγκλημα, τότε θα ήταν πολύ θετικό να μας ε, υποστήριζε και η κοινή γνώμη στις προσπάθειές μας. Να καταλάβει δηλαδή η κοινή γνώμη ότι θα μπορούσαν να είναι πολλά πράγματα καλύτερα τα νοσοκομεία, οι συντάξεις μας, τα συνταξιδοτικά ταμεία, αν δεν υπήρχαν αυτού του είδους υλοβιτούρες. Σας ευχαριστώ λοιπόν, αλλά φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Για να απαντήσω στον Μπίλι. Η κοινή γνώμη είναι με, μαζί μας, έτσι είπα. Γιατί η κοινή γνώμη θέλει διαφάνεια, θέλει. και γνωρίζει ότι στην κρίση υπάρχει μια εγκληματική διάσταση. Και οι εθνικές αρχές όμως και η κοινή γνώμη ίσως να μην έχουν καταλάβει το βαθμό στον οποίο υπάρχει σαπίλα και διαφθορά. Αυτή είναι που μας κρατάει άνεργους και φτωχούς και το ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος βέβαια και όλοι αναγκάζονται να πληρώνουν υψηλότερους φόρους από ό,τι θα έπρεπε. Και κάτι ακόμα που νομίζω ότι δύσκολα το εξηγούμε στους πολίτες μας είναι ότι είτε είναι υπέρ περισσότερης είτε λιγότερης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εφόσον είναι ότι πολλά από αυτά τα φαινόμενα δεν μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε ο καθένας μόνος του ή μικρή Πορτογαλία ή Ιρλανδία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα μικρή όλες είναι μικρές σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο γιατί θα αναγκαστούν αργά ή γρήγορα αν πολεμήσουν μόνες τους να εμπλακούν σε αυτά τα δε πολύ ευρεία δίκτυα ή αλλιώς θα αναγκαστούν να γίνουν και αυτές νέα, νέοι φορολογική παράδειση. Τα έχουμε δει αυτά και μέσα στην Ένωση. Ορισμένες χώρες ξεπλένουν χρήματα της ρωσικής ολιγαρχίας ή από την Αφρική. Έχουμε δει εταιρείες της Ένωσης να στηρίζουν δικτατορίες του τρίτου κόσμου. Επομένως δεν μπορεί καμία χώρα να τα καταπολεμήσει όλα αυτά μόνη της. Ευχαριστώ Ρουί, ναι, και επίσης ε, είναι πολύ σημαντικά τα όσα είπε ο Μπίλ στο βαθμό ότι εμείς πρέπει να κάνουμε την κοινή γνώμη και τους πολίτες να κατανοήσουν ότι αυτή η κρίση οικονομική κυρίως ε, προκλήθηκε όχι μόνο από την κακή συμπεριφορά των τραπεζών, αλλά και από την κακή συμπεριφορά μιας ε, πολιτικής και θεσμικής τάξης που δεν ε, μπόρεσε να σταματήσει αυτή τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος γιατί εμείς θα πρέπει να δώσουμε και κάποια αριθμητικά στοιχεία αλλά θα πρέπει να παγιώνονται από στοιχεία, να μιλούνται από στοιχεία αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Δηλαδή, ποια είναι η επίπτωση στην οικονομία και των 27 κρατών μελών της δράσης του οργανωμένου κλίματος. Ε, και εγώ ξέρω ότι οι πολίτες μας όταν ε, μάθουν τα στοιχεία αυτά θα αρχίσουν να φοβούνται γιατί το μόνο νούμερο που υπάρχει σήμερα έχει να κάνει με την Ιταλία και μπορώ να σας πω ότι δεν είναι πραγματικό νούμερο. Έχουμε ένα νούμερο που είναι σε μείωση γιατί αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι αυτό που έχει προκύψει από τις ερευνητικές δραστηριότητες αλλά πόσα ακόμη δεν γνωρίζουμε και είναι υπόγεια Ποιες είναι οι συναλλαγές ε, που όσο εμείς ε, μιλάμε υλοποιούνται από τη μαφία και το οργανωμένο έγκλημα και αυτό εις βάρος των Ευρωπαίων πολιτών και εις βάρος του πορτοφολιού των Ευρωπαίων πολιτών. Εγώ είμαι σίγουρη ότι όταν γνωστοποιηθούν όλα αυτά, κανένας πολίτης ε, δεν θα παραμείνει αδιάφορος. Το αντίθετο θα ζητήσει από τις κυβερνήσεις της Ένωσης να παρέμβουν, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Μπίλ αν ε, δεν υπήρχε αυτή η συνεχής πρόοδος από οικονομική, πολιτική, κοινωνική, θεσμική σκοπιά, τίποτα δεν αποκλείεται από το πόσο προχωρά σε αυτούς τους θεσμούς ε, το οργανωμένο έγκλημα, αλλά εγώ νομίζω ότι αν ε, δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο, νομίζω ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ε, αξιόλογο σύστημα υγείας και θα μπορούσαν ε, ε, όλοι να έχουν μία θέση εργασίας. Πρόκειται για κάποια νούμερα γιατί, κοιτάξτε, και το οργανωμένο έγκλημα θέτει ένα δικό του οικονομικό στόχο, αλλά η διαφθορά ποιε επιπτώσεις έχει στον οικονομικό ιστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θέλω να επενδυμίσω το νούμερο που έδωσε η κυρία Μάλστρομ ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Μιλούσε για 120 δισεκατομμύρια ευρώ για 27 χώρες. Όμως αυτά τα 100, από αυτά τα 120 μόνο τα 60 ε, έχουν εντοπιστεί στην Ιταλία. Εγώ όμως δεν νομίζω ότι η Ιταλία είναι η μόνη χώρα ε, στην οποία έχουμε δραστηριότητες σε τέτοιο βαθμό. Είναι πολύ χαμηλό αυτό το νούμερο. Μιλάμε για πάρα πολύ υψηλά νούμερα. Και εγώ είμαι πεπισμένη ότι τα κράτη-μέλη γνωρίζουν ποια είναι αυτά τα νούμερα, αλλά πολλές φορές μπορεί να φοβούνται να παραδεχτούν στους πολίτες τους ότι δεν μπόρεσαν ε, να καταπολεμήσουν το φαινόμενο. Γιατί, ε, κοιτάξτε, όλα αυτά που έχουν γίνει ε, για την καταπολέμηση των φαινόμενων αυτών δεν έγινε μία νυχτή. Ας θυμηθούμε πόσες φορές πήγαν οι Ιταλοί ερευνητές στη Γερμανία για να υποστηρίξουν πόσο αναγκαίο είναι να δοθεί ύψιστη προσοχή στα θέματα αυτά. Και πόσες ε, φορές οι δικαστές μας επέστρεψαν στην Ιταλία με αδιαχέρια γιατί η νομοθεσία στην ε, Γερμανία δεν προσφέρουν κάποιες συγκεκριμένε ε, δυνατότητες και κατόπιν όταν είχαμε την καταστροφή του Duisburg. Και τότε χύθηκε αίμα στους γερμανικούς δρόμους και υπήρχε φόβος ε, των Γερμανών πολιτών ε, ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί ε, οπουδήποτε με τέτοια επίθεση της μαφίας, τότε προσπάθησαν λοιπόν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Όμως η πραγματικότητα που αυτοί θεωρούσαν είναι πολύ μακρινή από το τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, εμείς πρέπει να υποστηρίξουμε το κάνουμε. Έχουμε πίσω μας μισή χρόνο ύπαρξης αυτής της Επιτροπής. Εμείς έχουμε ως στόχο να κάνουμε τα κράτη-μέλη να δουν την αναγκαιότητα να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα και με ένα νομοθετικό σύστημα να διορθώσουν την κατάσταση, να επανορθώσουν. Γιατί εγώ ειλικρινά και νομίζω ότι και εσείς πάρα πολλές φορές εδώ έχουμε ακούσει ερευνητές, ειδικού, δικαστές. Θα θυμάται τι είπε ο Μπερνάρ Φίγκερ, ο επικεφαλής ε, της αστυνομίας στο Βερολίνο, όταν είπε ότι εγώ θέλω και στη χώρα μου να υπάρχει ως αδίκημα η σύσταση σε μαφιόζικη συμμορία. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να φτάσει στην κυβέρνηση στη Γερμανία, στους γερμανούς πολιτικούς. Γιατί όταν μιλάμε για την οικονομία μιας χώρας, για τη σταθερή οικονομία, η σταθερή οικονομία αξιολογείται βάσει της διαφάνειας που υπάρχει στην οικονομία της χώρας αυτής. Ο κύριος Μποργκέτσιο. Ευχαριστώ. Θέλω να πω κάτι σε σχέση με όσα είπατε. Εγώ θα πρότεινα και με τη βοήθεια της γραμματείας να προσπαθήσουμε να βάλουμε αριθμητικά στοιχεία στην δική μου έκθεση για να έχει κάποια στοιχεία επαλήθευσης. Εγώ έχω κάποια στοιχεία του 2009 που δεν αναφέρονται και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, βεβαίω, λέει ο πρόεδρο, γιατί ο κύριο ε, στόχο, αν ε, θέλουμε να ψηφίσουμε την ε, προσοχή των Ευρωπαίων πολιτών, είναι να του κάνουμε να καταλάβουν τι συμβαίνει. Αναφέρθηκε και ο κύριο Νιούτον στο σκάνδαλο του Φίντου που τράβηξε την προσοχή όλων των πολιτών. βλέπουμε ότι και κάποια τμήματα της πολιτικής αλλά και των θεσμών ή έκλειναν τα μάτια, δεν ήθελαν να λάβουν δράση πολλές ε, φορές, όμως όχι μόνο ε, έκαναν ότι δεν έβλεπαν, αλλά ανακατεύτηκαν και όλες έβαλαν ε, τα βρώμικα χέρια τους σε αυτές τις υποθέσεις και σήμερα μας ε, προτείνονται ως επανάκια. Λοιπόν, αν ε, δεν υπάρχουν άλλες ε, παρεμβάσεις, να ολοκληρώσουμε εδώ. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9. Τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω τους συζητητές να παραμείνουν στην αίθουσα, ίσως να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Έρχεται και ένας ακόμη συνάδελφος για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Οι υπόλοιποι παρακαλώ να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί.